όμως για ένα καλύτερο μέλλον στην ευρωπαϊκή οικογένεια που ανήκουμε. Ευχαριστώ. Για όσους ανησυχούν θα πρέπει να καθησυχαστούν γιατί η Κομισιόν αντιπροσωπευόταν εδώ από τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για τον προπολογισμό. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν την συζήτηση αυτή αύριο με την, ψηφοφο... με την ψηφοφορία. Επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη είναι η κοινή συζήτηση περί της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε την έκθεση του κύριου Γκέρενς για το πρόγραμμα, της, το μέλλον μάλλον της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια ερώτηση προς την Επιτροπή 2015 Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη. Πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Γκέρενς. Monsieur le Président,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 Κύριε Πρόεδρε, γιατί να πρέπει να αλλάξει η πολιτική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί πλέον να μείνει ίδια γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει. Τη σήμερα ημέρα 7 φτωχοί στους 10 στον κόσμο δεν ζουν πλέον στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στις αναπτυσσόμενες αλλά στις αναδυόμενες χώρες. Η παγκοσμιοποίηση είναι αλήθεια, δημιουργεί σημαντικά πλούτη τα οποία ωστόσο δεν αγγίζουν τους πιο στερημένους. Αυτά όλα ε, προστίθεται, προστίθεται μια μεγάλη δημογραφική ανάπτυξη. 7 δισεκατομμύρια στόματα ε, που θα γίνουν 9 σε 20 χρόνια. Το ποσοστό οικονομική ανάπτυξη μια χώρα δεν ε, πραγματοποιείται παρά μόνο τη στιγμή που ξεπερνά το ποσοστό γεννητικότητα. Κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα το βάρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο θα μειώνεται διαρκώ, πράγμα που ορισμένοι ονομάζουν ε, στρατηγική παρακμή, αντίθετα από τι αναδυόμενε χώρε που ήδη έχουν, αποτελούν πολιτικού φορεί χωρί κανένα σύμπλεγμα. Ωστόσο, παραμένει το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτο παγκόσμιο φορέα όσον αφορά την δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια. Θέλει να παραμείνει πρώτη, αλλά και, καλύτερος, και καλύτερη σε αυτό το τομέα. Ορίστε κάποιες, ειδού κάποιοι προβληματισμοί τη Επιτροπή ανάπτυξη ώστε αυτό να ε, γίνει στο μέλλον. Η αναπτυξιακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί του πιο ευγενεί στόχου να προωθήσει την ανθρώπινη εξωπρέπεια, ριζώνοντα τη φτώχεια. Τίποτα λιγότερο. Η αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να προσανατολίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες των νοτίων εταίρων μας, σεβόμενοι τι επιλογέ τους. Θα πρέπει να εξυπηρετεί τους στοχούς χωρίς ε, ε, άλλες προσδοκίες και να σέβεται τις συμφωνίες του Συμβουλίου ε, της Κομισιόν και του Ευρωκοινοβουλίου. Προτείνουμε η Λέδη Άστον να, υπογράφει επίσης το, να υπογράψει επίσης το εν λόγω έγγραφο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την Ανάπτυξη, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία όσον αφορά την αναπτυξιακή πρόθεση της Ένωσης. Εμείς κάνουμε έκκληση προς όλους, ιδιωτικούς φορείς, πλούσια κράτη, φτωχά κράτη, πολυμερείς φορείς, ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες του σε θέματα ανάπτυξη. Γι' αυτό στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βούλησή της να διαφοροποιήσει τη βοήθειά της και να εξαλείψει από τον κατάλογο των δικαιούχων τη αναδυόμενης χώρας των οποίων η οικονομία διαρκώ ε, αναπτύσσεται. Η καταπολέμηση τη στόχη τη χώρα αυτές δεν πρέπει πλέον να, ε, να απόκειται στην διεθνή αλληλεγγύη αλλά στην εσωτερική τους πολιτική. Η Κομισιόν θα ήθελε αυτό να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο διαλόγου με τις χώρες αυτές και μέσω μια σταδιακής απόσυρσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, της βοήθειάς της προς αυτές. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ είναι υπέρ μιας καθολικής ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστό, εμείς τη στηρίζουμε αυτή την προσέγγιση. Ωστόσο, θα πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν προωθεί τη βελτίωση της ε, διαβίωσης των, φτωχο... των... Πιο... των φτωχότερων. Θα χρειαστεί να λεφθεί αυτό υπόψη στην προγραμματισμό της βοήθειας. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί τουλάχιστον 20% βοήθεια στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως αυτές ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη μέσα στους στόχους της χιλιετίας για την ανάπτυξη. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει δεν να είναι και συνεπής. Συνέπεια σημαίνει ε, άλλα τμήματα εκτός από την ανάπτυξη να πάψουν οποιαδήποτε διάβημα που μπορεί μέσω της δράσης τους να καταστρέψει τα όσα φτιάχτηκαν χάρη στην αναπτυξιακή βοήθεια. Θα πρέπει τα 27 κρατημέλη να λειτουργούν μαζί έτσι ώστε όταν θα είναι 28 μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την, εξωτερική, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να ανταποκρίνονται στον συντονισμό που προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ο εισηγητής σας θεωρεί ότι ο διάλογος μεταξύ των 28 είναι, δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Όσον αφορά την υπουργική συμμετοχή στη συνεδρία του Συμβουλίου και όσον αφορά το περιορισμένο χρόνο που αφιερώνεται σε αυτό το θέμα. Θεωρώ πως είναι απαραίτητο η λήψη αποφάσεων να τις λήψεις αποφάσεων να προηγείται η οργάνωση ενός ε, μιας συνένεσης γύρω από τις βασικές, ε, τα βασικά πολιτικά θέματα, τα στρατηγικά θέματα που καθορίζουν την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης. Ένα ανεξάρτητο δηλαδή κύτταρο προβληματισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα δώσει προστιθέμενη αξία σε σχέση με τους εθνικούς ε, οργανισμούς που ήδη υπάρχουν για να ανταποκριθούμε καλύτερα στα, στις μεγάλες προκλήσεις της ανάπτυξης. Και δεν χρειάζεται να σας αναφέρω όλες τις λεπτομέρειες. Ε, θα τα βρείτε όλα αυτά στην έκθεσή μου. Γραπτά. Το γνωρίζουμε ότι δεν αναπτύσσουμε αρκετά την ανάπτυξη στη δημόσια συζήτηση για να διορθωθεί αυτό και αυτό είναι και το θέμα της προφορικής μου ερώτησης. Ε, μαζί με την έκθεση την υπέβαλα Θέλουμε το Ευρωκοινοβούλιο να, να εκφραστεί υπέρ της πρότασής μας ώστε το 2015 να οριστεί ως έτος, Ευρωπαϊκό έτος της ανάπτυξης. Αυτό στηρίζεται και από τον κύριο, τον φίλο ε, Μπέρμαν, τον συνάδελφο Μπούλα και την Εύα Ζολή. Γιατί υπεύθυνη ανάπτυξη, διότι η αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας δεν θα επιτευχθούν εάν τα κράτη με μέσο εισόδημα ζουν, στα οποία ζουν 7 φτωχοί από τους 10 δεν αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η υπεύθυνη ανάπτυξη μας οδηγεί στο να σκεφτούμε ξανά κάποιες μεθόδους μας. Αν θέλουμε να, να έχουμε βάρος το 2015 δεν νομίζω πως είναι πια πρόημο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουλάν έχει τώρα το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον Σαλ Γκορέντς για την εξαιρετική του έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει πάνω από το 50% της αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο. Ε, ακόμα και μετά το... Όμως μέχρι το 2015 ε, παρόλο ότι θα έχουμε πετύχει κάποιους από τους στόχους μας, ε, ε, δεν είμαστε τόσο πολύ συνεπείς σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική, την εμπορική μας πολιτική, την αγροτική μας πολιτική. Η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένες με και μετρήσιμες δεσμεύσεις και με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, βραχυπρόθεσμο. Ε, ο οικονομικός ανταγωνισμός, η ισχύ των αναδυόμενων οικονομιών, η κλιματική αλλαγή κλπ. μας επιβάλλουν καινούριε προτεραιότητε. Ασφάλεια των τροφίμων, πρόσβαση σε ενεργειακού πόρου και πρόσβαση σε υπηρεσίε υγεία. Σαφές ότι, είναι σαφές ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή συνένεση, αλλά θα πρέπει να ξαναδούμε το θεσμικό μας και το διεθνές σύστημα σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό τομέα, εμπνεόμενοι από οργανισμούς που ήδη λειτουργούν σωστά, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου για παράδειγμα. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στους ε, πολίτες μας ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δεν αποτελεί ε, ένα ε, φιλανθρωπία είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τις αγορές που ανοίγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις αναδυόμενες αγορές όπως η Κίνα, η Βρεσλία, η Ινδία. Επίσης θα πρέπει να δούμε την ε, ε, γεωστρατηγική μας πολιτική ε, τα τελευταία χρόνια, γιατί πλέον οι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν μεγεθυνθεί πολύ. Θα πρέπει λοιπόν και αυτές οι χώρες να συνεισφέρουν στη διεθνή σκηνή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει μια υπεύθυνη αντιξιακή βοήθεια σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Το 2015 ε, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ξαναδούμε την και μας βοήθεια, να μην τη βλέπουμε μόνο ως οικονομική βοήθεια, αλλά ως μια ε, υποστήριξη της ε, υπεύθυνα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η Επιτροπή Δευτεριών και οι η ΟΚΕ έχουν ζητήσει το 2015 να είναι έτος ανάπτυξης και συμφωνώ. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος. Ο κύριος Μπέρμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμπληρώνω την εξαιρετική παρουσίαση και έκθεση ε, του κύριου Γκιόρες και να κάνω τρία σχόλια. Η ατζέντα για την αλλαγή λέει σωστά ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη σύνδεση μεταξύ της ε, αναπτυξιακής πολιτικής και της επίγουσας βοήθειας. Στη χώρα μου, στις κάτω χώρες, ε, κάποιοι ζητούν να περιοριστούμε στην επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι παράλογο. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τη φτώχεια και τους ε, ε, πρόσφυγες. Κοιτάξτε τι γίνεται στο Μαλί. Αυτά είναι τροφή για τους φανατικούς μουσουλμάνους που πρεσβεύουν τη Σαρία και είναι αιστεία ανάφλεξη, ένα Αφγανιστάν κοντά στα σύνορά μας, στο Βόρειο Μαλί. Για να ξεφύγουμε από εκεί, να δούμε τι γίνεται στη Λατινική Αμερική ε, όλο και περισσότεροι εγκληματίες ε, έχουν ε, πρόσβαση στα λιμάνια της Γουινέας Μπισάου στη Δυτική Αφρική και μέσω της Σαχάρα φτάνουν τα ναρκωτικά στην Ευρώπη. Για να βοηθήσουμε το Μαλί λοιπόν δεν θα βοηθήσουμε μόνο τη χώρα αλλά και τους του ΑΡΕΚ και γενικότερα την ειρήνη στην περιοχή. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά το 2015 να έχουν όλη την ευκαιρία να βγουν από τη φτώχεια. Γίνεται ε, λοιπόν δημόσια συζήτηση και χρειάζεται αυτή. Καλό θα ήταν λοιπόν ε, να προχωρήσουμε. ένα καλό που η Ένωση ε, θέλει το 2015 είναι ευρωπαϊκό έτος για την ανάπτυξη. Ελπίζω να μας βοηθήσει ο κύριος Πίμπαλξ ε, να πετύχει αυτή η προσπάθεια. Χωρίς ανοιχτή δημοκρατία οι ίσες ευκαιρίες είναι χήμερα. Όσο δεν έχουν φωνή οι πιο φτωχοί στις δικές τους πρωτεύουσες τόσο δεν θα γίνονται πουθενά ακουστοί. Θα πρέπει λοιπόν να ακούγονται οι φτωχότεροι των φτωχών στα τοπικά κοινοβούλια, στα περιφερειακά, σε κοινωνικές οργανώσεις σε ΜΚΟ, σε οργανώσεις μειονοτήτων ή γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το επιλέγει και το υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω και το Συμβούλιο να ευθυγραμμιστεί σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Και τώρα θα ακούσουμε τη φωνή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, διαστόματος του κυρίου Πίμπαλξ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, νομίζω ότι καταρχά θα πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Γκέρεν για την εξαιρετική του έκθεση, αλλά και για τη συζήτηση που ξεκίνησε εδώ. Ε, σίγουρα αυτό χρειάζεται περισσότερη προσοχή, ε, αλλά χαίρομαι και ευχαριστώ την Επιτροπή Αναπτυξιακή συνεργασία που είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψει για την αναπτυξιακή πολιτική. Γιατί η αναπτυξιακή συνεργασία είναι από τι πιο περίπλοκες πολιτικέ στην Ένωση γιατί έχει ρόλο όχι μόνο την υποστήριξη των χωρών για την ανάπτυξή τους, αλλά αφορά και τη δράση μας σε άλλους τομείς πολιτικής. Επίσης είναι γεγονός αυτό που είπε ο κύριος Μπουλάν, ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε την αναπτυξιακή πολιτική όχι μόνο από το πρίσμα της αλληλεγγύης. Η αλληλεγγύη είναι σίγουρα ένα τμήμα της, αλλά είναι και επένδυση για την ασφάλεια των πολιτών μας και για την ευημερία των πολιτών μας. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολιτικές εγκάρσεις που ενισχύουν την Ένωση, η αναπτυξιακή πολιτική, εάν γίνουν με το σωστό τρόπο και αν γίνουν με λάθος τρόπο αποδυναμώνουν την Ένωση. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στον κόσμο προς το καλύτερο και τώρα έχουμε μοναδική ευκαιρία στη ζωή μας, όχι μόνο να προχωρήσουμε ε, και ε, να εξαλείψουμε τη φτώχεια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το κάνουμε και η Ένωση θεωρείται αξιόπιστος εταίρος. Τηρούμε πάντα τις υποσχέσεις μας, καμιά φορά με βραδύτητα, αλλά είμαστε πραγματικά ειλικρινεί στην προσέγγισή μας. Δεν έχουμε ιστεροβουλίες. Είμαστε ειλικρινεί και θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες να ορθοποδούν. Έτσι λοιπόν, θέλουμε να ακολουθήσουμε μια πιο στρατηγική ε, κατεύθυνση. Για να γίνει αυτό χρειάζεται κανείς να κάνει επιλογές. Και η αφετηρία μας είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, και η προσέγγιση αυτή ε, σημαίνει ότι δεν ε, διαχωρίζεται αυτή η πολιτική από την πολιτική για την υγεία, για την παιδεία, για τη στέγαση και για άλλα στοιχεία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συνοχή παντού και χαίρομαι πάρα πολύ που η έκθεση του κυρίου Σαρλ Γκέρενς ε, τα βλέπει όλα αυτά θετικά για μια υφόρο ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Ε, επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε να λέμε τι θέλουν οι εταίροι μας. Όχι γρήγορη ανάπτυξη του ΑΕΠ ε, με διψήφιους αριθμούς ή τριψήφιους αριθμούς. Δεν σημαίνει πάντα η αύξηση, η μεγένθηση του ΑΕΠ, ε, ανάπτυξη ενός λαού και μιας οικονομίας. Και αυτό σημαίνει κοινωνική ένταξη, κοινωνική προστασία είναι πολύ σημαντική, αλλά και η βιωσιμότητα και η αεφορία. Δεν αρκεί να έχει υψηλού ρυθμούς ανάπτυξης μια χώρα και μετά ε, να καταστρέφει το περιβάλλον της. Τι νόημα έχει αυτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση. Και δύο ζητήματα εδώ έχουν μεγάλη σημασία. Το ένα είναι πρόσβαση σε αηφόρες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αλλά και για την οικονομική μεγέθυνση. Αν δεν γίνει αυτό, ε, βλέπουμε σε κάποιες χώρες που κυριαρχεί η βιομηχανία και η ενέργεια από άνθρακα και κάποιες άλλες ε, υπολείπονται. Και το άλλο είναι η επισητιστική ασφάλεια. Δηλαδή, δεν θα έχουμε μόνο ανθρωπιστική βοήθεια. Το είπε και ο κύριο Μπέρμαν. Όλο και περισσότερο έχουμε θεομηνίε φυσικέ καταστροφέ και πιο ακριβέ. Και δεν βοηθάει απλώ να σώσει μια ζωή, μια συγκεκριμένη στιγμή τη θεομηνία. Θα πρέπει ο κόσμο να βοηθηθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του. Γι' αυτό και με τη συνάδελφο ε, Κρυσταλίνα Γεώργεβα και με τους ε, Βραζιλιάνους ε, συνεργαζόμαστε για να εξοικονομούμε χρήματα και σε κάποια στιγμή στην ανάπτυξη να βοηθήσουμε η ε, Βραζιλία είναι σε θέση να αναλάβει μόνη της ε, τώρα τις ε, τύχες της. Θα ήθελα να σχολιάσω κάτι που είπε ο Σαρλ για το διάλογο με τα κράτη-μέλη. Έχουμε προχωρήσει το Συμβούλιο Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Μπορεί να μην είναι το πιο σημαντικό αυτό, αλλά το Μάιο είχαμε μια ολόκληρη ημέρα αφιερωμένη σε αυτό το Συμβούλιο, παρουσία της κυρίας Άστον ε, ξέρουμε ότι είπατε εκπρόσωπος που είναι πάρα πολύ απεισχολημένη, αφιέρωσε ολόκληρη ημέρα ε, στο Συμβούλιο Υπουργών Ανάπτυξης. Καταλαβαίνετε πόση σημασία έχει αυτό. Συμμετέχουν πλήρως τα κράτη-μέλη. Και ένα άλλο ορόσημο είναι το κοινό πρόγραμμα. Και χαίρομαι τώρα που έχουμε και από τη Γαλλία υποστήριξη. Ο Υπουργός Καλφάν θα βοηθήσει και δεν είναι μια προσπάθεια που κάνει μόνη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να εστερνίζονται πλήρως αυτή την πολιτική. Και ένα τελευταίο, χωρίς να είναι αυτό το λιγότερο σημαντικό, για τη διεθνή συμμετοχή. Καμιά φορά λέμε ότι μας παρεξηγούν ε, γιατί τώρα έχουμε μια ιστορική ευκαιρία σε αυτή τη διαδικασία για το 2015 και επέκεινα. Ε, ε, οι στόχοι της χιλιετίας ε, έχουν αλλάξει τη ζωή ε, των ανθρώπων και το 2015 εκπνέουν. Ολοκληρώνεται αυτή η προσπάθεια που τη γνωρίζει πολλοί κόσμος και θα πρέπει από εκεί να ε, κινήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως και να είναι σημαντικός ε, πρωταγωνιστής. Αυτά. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έτος 2015 για την αναπτυξιακή συνεργασία και μάλιστα ορόσημο θα το χαρακτήριζα. Ε, γι' αυτά, λοιπόν, για αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι η διοργάνωση ενός Ευρωπαϊκού έτους για την ανάπτυξη το 2015 θα είναι και επίκαιρο και εύστοχο ε, γεγονός σε επίπεδο ένωσης θα είναι καταλήτης και θα συγκεντρώσει την προσοχή και της κοινή γνώμης αλλά και εκείνων που παίρνουν τις αποφάσεις για θέματα ανάπτυξης και ιδιαίτερα για τους στόχους της ανάπτυξης μετά το 2015. Σημειώνω και την υποστήριξη ε, της Επιτροπής των Περιφερειών και ε, του Προέδρου του Κοινοβουλίου. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τι συνέπειες θα έχει αυτό και τα υπόλοιπα οργανωτικά θα πρέπει επίσης να κινητοποιήσουμε ανθρωπίνους πόρους επαρκής για να βεβαιωθούμε ότι θα στεφθεί με πλήρη επιτυχία μια τόσο μεγάλη εκστρατεία. Όλα αυτά τα βλέπουμε θετικά, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να βεβαιωθούμε ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να δώσουμε και αποτελέσματα πριν δρομολογήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Θα επανέλθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με λεπτομερείς προτάσεις, ε, ακολουθώντας τη κανονική διαδικασία για ε, τον καθορισμό ενός ευρωπαϊκού έτους. Και ε, προσβλέπω και υπολογίζω και στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου ως δημοσιονομική αρχή για να έχουμε επαρκείς οικονομικούς πόρους, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα έχει επιτυχία μια τέτοια διοργάνωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much, Mr. Commissioner. In the name of the European... Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Για το Ευρωπαϊκό Λογικό Κόμμα ο κύριος Κάτσμαρέκ για ένα μισή λεπτό. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Η Επιτροπή Ανάπτυξης αποφάσισε να ασχοληθεί με την έκθεση για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια, γιατί βεβαίως μιλάμε για τα βασικά ζητήματα της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Γκέρεντς που ασχολήθηκε με αυτή τη σημαντική πρόκληση και συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να δούμε το ζήτημα της ε, βελτίωσης ε, των συστημάτων. Όταν ε, τα λεφτά σπανίζουν πρέπει να μετράμε κάθε ευρώ που δίνουμε. Και βεβαίως πρέπει να εξυγχρονιστεί και η αναπτυξιακή πολιτική γιατί ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Οπότε έτσι πρέπει να αλλάξουμε και εμείς. Ελπίζω λοιπόν να επιτύχει αυτή η αλλαγή. Η έννοια αυτή της ε, ολοκληρωμένης ανάπτυξης συμφιλιώνει την οικονομική ανάπτυξη με τις νέες εξελίξεις στον ε, κοινωνικό τομέα. Πρόκειται για κάτι το καθαρά ευρωπαϊκό, η κοινωνική οικονομία της αγοράς. Οπότε βλέπουμε ποιος είναι ο στόχος, δηλαδή η αντιμετώπιση της ε, φτώχειας. Πρέπει λοιπόν η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική να είναι ολοκληρωμένη και είμαι σίγουρος πως ε, με την έκθεση αυτή ερχόμαστε και κοντά στο να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σας ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Κόρτες Λάστρα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να συγχαρώ τον ε, κύριο Γκέρενς για αυτή την έκθεση. Παίρνει μια ισχυρή θέση που οριοθετεί την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης. Και αυτό μέσα σε ένα πλαίσιο περικοπών σε όλη την αναπτυξιακή βοήθεια στην Ένωση. Και αυτό μέσα στα πλαίσια των στόχων της χιλιετίας του 2015 το μήνυμα που θα υποστηρίξει το Κοινοβούλιο αύριο είναι σημαντικό. Ναι μεν, οι καιροί αλλάζουν, οι συγκυρίες αράζουν, αλλά οι Ευρωπαίοι εμείς πάντα ποντάρουμε για την ανάπτυξη, τη συνεργασία, για την αλληλεγγύη. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το σώμα θέλει αηφόρο ανάπτυξη, ανακατανομή του πλούτου και κοινωνική δικαιοσύνη με χρηματοδότηση στο ύψος των προκλήσεων. Το 70% των φτωχών στον υπόλοιπο κόσμο δεν θα πρέπει να τύχει περικοπών βοηθείας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε σημαντικά τη συμμετοχή μας σε τριγωνικές συμφωνίες συνεργασίας και δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στο ΑΕΠ μιας χώρας για να ορίσουμε το ύψος της βοήθειας αλλά θα πρέπει να Μπούμε και το βιωτικό επίπεδο. Ζητούμε να δοθεί φρόνημα λογικά η ευρωπαϊκή βοήθεια η οποία έχει προστιθέμενη αξία και είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σαρτζεντίνη, εξ ονόματος των Πρασίνων, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Κέρνς για την πολύ καλή του έκθεση. Αλλά αυτό το οποίο μου φαίνεται ένα πρόβλημα είναι πως σε καιρούς οικονομικής κρίσης θα προσαρμόσουμε το όραμα της αναπτυξιακής πολιτικής. Και αυτό θα ήταν καλό εάν ήμασταν έξυπνοι, εάν λέγαμε πως η αφετηρία μας είναι η συνοχή της πολιτικής και πως θα ασκήσουμε πίεση και για το εμπόριο και για τις επενδύσεις. Αλλά εάν δεν το κάνουμε και κοιτάμε μόνο πόσο μπορούμε να βάλουμε στα επίσημα ταμεία μας αναπτυξιακής βοήθειας, τότε φοβάμαι κύριε Πίμπαλξ πώς ασχολούμαστε με το να δίνουμε επιχειρήματα στην αντίπαλη πλευρά. Δηλαδή, μπορείτε πιο αποτελεσματικά, άρα μπορείτε με λιγότερα λεφτά. Το βλέπω και στη χώρα μου, όπου είχαμε μείωση του αναπτυξιακού προϋπολογισμού από 0,8 στο 0,7 του ΑΕΠ. Οπότε το ερώτημά μου κύριε επίβαλξη, είναι πότε πραγματικά θα είμαστε έξυπνοι και τίμοι σε αυτές τις επενδύσεις τις οποίες κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την Γκουε ο κύριος Όμαρτζε. Για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θα επιμείνω σε ένα σημείο από όλα όσα συζητήσαμε, την Αφρική. Στην Αφρικανική Ήπειρο τίθενται όλα αυτά τα ζητήματα με τον πιο βαρύ τρόπο. Και στην Αφρική βρίσκονται και μετα... βρίσκεται και το μεγαλύτερο δυναμικό. Το Η δημογραφική ανάπτυξη στηρίζει αυτήν, αυτό το διπλό πρόσωπο. Ο πληθυσμός της Αφρική σε μερικά χρόνια θα διπλασιαστεί. Μπορεί λοιπόν αυτή η Αφρική να γίνει ένας μοχλός πρόοδου και ανθρώπινης ανάπτυξης ή λόγω της ανικανότητάς μας εγκρίζωσης της παινίας η Αφρική θα καταστεί ένας πόλος αποσταθεροποίησης του κόσμου. Δεν πρόκειται για μία απλή πολιτική ε, φιλανθρωπίας μια πραγματική αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να αποτελεί επένδυση για το μέλλον που θα υποστηρίζει μια μεγάλη φιλοδοξία για την ίδια την Αφρική αλλά και για την δική μας την Ήπειρο. Η μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται και η Κίνα εξάλλου το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά. Και η ειρήνη στον κόσμο εξαρτάται επίσης πολύ από αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Μίτσελ για μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω τον Charles Γκόρεντς και τον ε, Επίτροπο για την παρουσίασή του. Τρία σύντομα σημεία. Πρώτον, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον ε, οι οικονομίες των αναπτυγμένων χωρών θα μπορούν να αναπτυχθούν και αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσει να βοηθήσουμε τον ιδιωτικό τομέα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε, να εμπλακούμε και να έρθουμε σε επαφή με άλλους πολιτικούς για να το συμπεριλάβουν και αυτοί. Αυτό θα δώσει στους ανθρώπους το αίσθημα ότι τους ανήκει αυτή η εξέλιξη και θα έχουν μια αίσθηση του μέλλοντος. Επίσης πρέπει να ασχοληθούμε με αυτή τη συνεκτική πολιτική. Δηλαδή η Κομισιόν αναφέρθηκε σε μεγάλες εξοικονομήσεις σε περίπτωση που είναι συνεκτική αυτή η πολιτική και θα πρέπει με κάποιο τρόπο το Εθνικό αυτό Κοινοβούλιο αυτό σε συνομιλία με τα Εθνικά Κοινοβούλια να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσει την πενεπιρροή του για να το πετύχει αυτό ώστε να ξεπεράσουμε τους διστακτικούς υπουργούς, το Συμβούλιο Υπουργών οι οποίοι θέλουν να τα κρατήσουν σταματήσουν όλα για τους αυτούς τους και επίσης ο Υπουργός, ο Επίτροπος παρέμεινε σε μια εκδήλωση για τα δύο φύλλα. Υπάρχουν εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο που λείπουν, εξαφανίζονται λόγω των αμβλώσεων και δεν πρέπει αυτό να το ξεπεράσουμε. Δεν... Και αυτό πρέπει να το κάνουμε ζήτημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. The next speaker uh, η κυρία Στρίφλαρ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Γκέρενς για αυτήν την εξαιρετική έκθεση. Και λόγω της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης σήμερα που είναι δύσκολη είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να περιφρουρούμε το πώς ξοδεύεται αυτή η βοήθεια για να μας δίνει και τα καλύτερα αποτελέσματα. Πρέπει να έχουμε στοχευμένους, στο, ε, στοχευμένες παρεμβάσεις εκεί όπου υπάρχει και μεγαλύτερη ανάγκη. Θα πρέπει να έχουμε μία διαφοροποιημένη αντίληψη για τις εφαρμοστικές λεπτομέρειες της βοήθειας. Θα έπρεπε να βοηθήσουμε την γεωργία κυρίως και αυτό ενισχύοντας τις τοπικές πρακτικές, τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό η Κομισιόν να στοχεύσει τη βοήθειά της στην, στο γεωργικό τομέα, στην διατροφή στη, και όλα αυτά στη φάση της περίοδου 2014-2020 να, η καταπολέμηση της πενίας, η αποτελεσματική καταπολέμηση της ε, παινίας χρειάζεται συνέργεια μεταξύ ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας που αποτελούν απαράβατο όρο για να καταπολεμήσουν την απαγοήτευση και να ξεκινήσουν ε, τη διαδικασία της αηφόρου ανάπτυξης. Θα έλεγα λοιπόν έτος της ανάπτυξης ναι για την αηφόρου ανάπτυξη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Φύσασα Ξέλα για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Γκιόρενς για την εξαιρετική έκθεση. Το χρονοδιάγραμμα αλλαγής αποτελεί ένα φύλλο ε, για την αναζήτηση καλύτερης ποιότητας της ε, αναπτυξιακής βοήθειας και αυτό υπό το φως των αλλαγών που έχουμε στη νέα παγκόσμια τάξη, την ε, γέννηση νέων πρωταγωνιστών παγκοσμίω και επίσης τον φορολογικό ανταγωνισμό που μας οδηγεί στην τωρινή κατάσταση. Ε, θέλουμε η παινία να αποτελεί, η φτώχεια να αποτελεί ένα βασικό κριτήριο διαφοροποίησης ε, κριτηρίων επιλογής. Λυπόμαστε όμως που το ΑΕΠ αποτελεί κριτήριο επιλογής. Το 70% όσων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στον κόσμο ζουν σε χώρες με, μέσα, ε, με μέσο εισόδημα. Πέρα δηλαδή από το επίπεδο πλούτου της χώρας θα πρέπει να έχουμε και άλλα στοιχεία για κριτήριο, δηλαδή ε, ανάπτυξη ε, ανθρωπίνων πόρων, θα ε, συνοχή μέσα στη χώρα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε πόλους συνεργασίας νότος-νότος ή τριγωνικές συμφωνίες συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μπάγκο. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ γράφτηκα για το ένα λεπτό. Με συγχωρείτε, αυτό το όνομά μου έδωσαν η κυρία Καστίγιο. Thank you, Um, I'm speaking here as well. Ευχαριστώ και εκπροσωπώ τον ε, κύριο Κάσμαν, ο οποίος είναι σκιώδης ηγητής για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και άργησε. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον συγητή για την εξαιρετική έκθεση και την ε, Κομισιόν ε, για την ε, εμπλοκή του στη σύνταξη της έκθεσης. Η έκθεση αυτή θεωρούμε έχει επιτύχει μια ισορροπημένη προσέγγιση στην ανάπτυξη. Καλωσορίζουμε την ε, πιο έντονη διατύπωση για την δικαιότερη κατανομή του πλούτου και ιδιαίτερα τη έμφαση που δίνεται στην αϊφόρο ανάπτυξη για όλους. Όσον αφορά την ε, διαφοροποίηση, τώρα καλωσορίζουμε την έντονη διατύπωση που υπάρχει για τον πολιτικό διάλογο, για την εξάλληψη της στόχιας ε, μέσω της εσωτερικής αλληλεγγύης με χρηματοδότηση και από τη δική τους πλευρά. Όμως δεν μπορούμε να κόψουμε απότομα τη χρηματοδότηση, ειδικά όσον αφορά τις χώρες της λεγόμενες μέσου εισοδήματος, ειδικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό. Πρέπει να υπάρχει ένας οδικός χάρτης ή μια στρατηγική εξόδου ειδικά όσον αφορά τις μικρότερες χώρες. Οι χώρες αυτές ε, είναι πιο ευάλωτες. Και πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κριστίνα Όριαν κατόπιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας τομέας ο οποίος συνδέεται άμεσα με την ΚΕΠΑ τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτική αλληλείας και κλίματος, στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας κτλ. Όμως, όπως σωστά επισήμανε ο εισηγητής, ο πολιτικός διάλογος μεταξύ διεθνών φορέων, αλλά και η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, κομισιών και της ε, σχετικής υπηρεσία δεν είναι ακόμα πολύ οργανωμένη. Το να υπάρχει λοιπόν συνοχή μεταξύ των διαφόρων φορέων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών πρέπει να είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν. Οπότε εγώ θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Επίτροπο να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης να επισημάνω πως όταν μιλάμε για αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να σκεφτούμαστε πολύ περισσότερες χώρες από τις χώρες ΑΚΕ. Έχει χρησιμοποιηθεί το μέσο, παραδείγματο χάρη αυτό, για να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη στην Ουκρανία και στον Νότιο Κάυκασο. Σας ευχαριστώ, κύριο Φερέιρα. Η αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης ουσιαστικά στερείται βασικών στοιχείων. Δεν έχει επαρκείς πόρους στο ύψος των στόχων της και των διεθνών συμφωνιών που έχει συνάψει στα πλαίσια του ΟΗΕ. Λείπουνε τα μέσα εκείνα για την χορήγηση βοήθειας που να ενισχύει την εθνική κυριαρχία ορισμένων χωρών. Δεν υπάρχει αυτός ο συνδυασμένος μηχανισμός ε, ο οποίος παράλληλα με τη βοήθεια στοχεύει και στην πρόβλεψη. Σχετικά με την ευκυβερνησία, οι πολιτικές πρακτικές σε πολλούς ε, τομείς όπως είναι η φορολογία, η δικαιοσύνη κτλ. Πολιτικές οι οποίες θα έπρεπε να αποτελούν de facto επιλογή των αναπτυσσομένων χωρών λαμβάνοντας υπόψη τις δικές τους ιδιομορφίες και όχι να τους εξάγουμε τα δικά μας μοντέλα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις τομιακές πολιτικές και την έλλειψη σύνοχης αυτών των πολιτικών με την ανάπτυξη. Ο κύριος Κέλλη. Uh, Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και δικαιολογημένα να είναι περήφανη για τη συνεισφορά της στην αναπτυξιακή βοήθεια εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτό υποθέτω ότι έχει και αναγνωριστεί στο γεγονός ότι της απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Καταρχήν για την αναπτυξιακή βοήθεια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ειρήνη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι γελιοποίησαν αυτή την απονομία, αλλά περισσότεροι από εμά μπορεί να αισθανθούμε μεγάλη περηφάνεια αυτό που έχουμε πετύχει και θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε στο, εσωτερικό να δημιουργούμε και να διατηρούμε την ειρήνη αλλά και στο εξωτερικό μέσω τη αναπτυξιακή βοήθεια και ιδιαίτερω να βοηθάμε τι χώρε να έχουν ειρήνη και βιωσιμότητα μέσω τη ανάπτυξη των οικονομιών του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τέλο, σε σχέση με αυτό που είπε ο Συνάδελφο Φύση είναι πολύ σημαντικό. Το ΑΕΠ δεν θα πρέπει να είναι ο κατά τη την αξιολόγηση των κρατών και των τόπων στους οποίους μπορούμε να επενδύσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κύριος Μπρόντς είναι το επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Η έκθεση αναφέρεται στην εντυπωσιακή ανάπτυξη της Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας. Αντί εντυπωσιακή, εγώ θα έλεγα απειλητική για τον μεταποιητικό ε, τομέα της Ευρώπης και κυρίως της χώρας μου, του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έκφραση εκφράζει έκθεση, έκπληξη που δεν μπόρεσαν οι χώρες αυτές να μειώσουν τη φτώχεια τους. Αλλά θα έλεγα ότι πάνω στη φτώχεια τους, για να μην πω στις συνθήκες ε, ε, δουλείας στην εργασία, στη αυτή ανάπτυξη θα πρέπει να μην τους χορηγείται μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή βοήθεια. Μόνο μασοπρόθεσμα, εν μεταξύ άμεσα καταστρέφουν το δικό μας τομέα. Η παγκοσμιοποίηση επίσης επενείται στην έκθεση υπό την έννοια ότι μειώνει τις ανισότητες μεταξύ των χωρών. Δηλαδή, οι αναδυόμενες χώρες γίνονται πλουσιότερες σε βάρος κάποιων από τους δικούς μας εργαζομένους. Όμως, οι ανισότητες εντός των χωρών αυξάνονται, καθώς οι εργαζόμενοι στα κράτη-μέλη πηγαίνουν στην ανεργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Τιρλιάν. Ε, ε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ατζέντα που προτείνει η Κομισιόν δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Το βασικό είναι η εφαρμογή των διαφόρων διαφοροποίησεων. Θέλει η Κομισιόν από το 2014 η επιλογή των χωρών που θα, στις οποίες επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ανάπτυξη να βασίζεται στο μηχανιστικό στοιχείο του ΕΠ. Και όπως το θύμισε και η κυρία Άστον, όλα αυτά τα ζητήματα δεν είναι λογιστικού χαρακτήρα. Χρειάζεται πολιτική συζήτηση για τις προτεραιότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό φυσικά δεν συμβαδίζει και με το πνεύμα του κοτονού. Οι χώρες ΑΚΕ που είχαν θετικά οικονομικά αποτελέσματα θα πρέπει να ενθαρρυνθούν στη μεταβασή τους σε μια πιο αηφόρα ανάπτυξη. Μπόρεσαν να εγγυθούν την ανάπτυξη αυτές οι χώρες μέσα από μια σωστή πολιτική και ευκυβερνησία. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο τώρα. Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Θα μου επιτρέψετε να διατρέξω γρήγορα τα σημαντικότερα για τον κύριο Κατσμάρεκ. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να γίνει καταλήτης η βοήθεια για να επιτύχουν τα αποτελέσματα αυτά μαζί με τους στόχους της ε, χιλιετίας ε, για να έχουμε ακόμη ισχυρότερη αλλαγή και θα έλεγα οπωσδήποτε πως η πρωτοβουσία η πρωτοβουλία Φάρα αφορούσε τις εξορρυκτικές δραστηριότητες που πρότεινε ο συνάδελφος ε, ο κύριος Μπαρνιέ. Εάν το εκμεταλλευτούμε αυτό μπορούμε να έχουμε ουσιαστική αλλαγή και σας ευχαριστώ που το υποστηρίσατε. Για τον ε, κύριο Ρικάρδο Κόρτες. Ε, για τη διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση δεν είναι μια φιλοδοξία και αυτός σκοπός. Ε, είναι η πραγματικότητα, αλλά κρατάμε νέα μέσα αναπτυξιακής συνεργασίας τα οποία θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε με τις ε, χώρες ε, εταίρους αλλά βεβαίω με κάποιες χώρες θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική γιατί το οικονομικό του επίπεδο και το μέγεθός τους απαιτούν άλλου τύπου συνεργασία για την κυρία Σαρτζεντίνη επενδύουμε επενδύουμε και σε αυτή την περίοδο βεβαίως ε, με βάση την ατζέντα για αλλαγή. Για τον κύριο Αμερτζή η Αφρική είναι πρώτη προτεραιότητα γιατί θα μπορούσε να γίνει μία ήπειρος ευημερία ή πλήρους καταστροφής. Οπότε πιστεύω πως η εμπλοκή μας στην Αφρική έχει κρίσιμη σημασία γιατί κανένας άλλος δεν θα στηρίξει τις αφρικανικές χώρες ε, για να επιτύχουν την ε, ευημερία και θεωρώ και ξέρω από τις επαφές μου πως θέλουν την Ευρώπη και κοιτούν προς την Ευρώπη όχι μόνο για λεφτά αλλά και για ενθάρρυνση και ανάπτυξη και εάν το εκμεταλλευτούμε αυτό θεωρώ πως η Αφρική θα αποτελέσει κινητήρα της ανάπτυξης στον πλανήτη και όχι μια ήπειρος με ανασφάλιση για τον κύριο Μίτσελ για αυτά τα οποία είπε Μα αυτό το γνωρίζουμε και από τον ιδιωτικό τομέα γιατί έτσι ενισχύονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, γιατί αν μιλάμε μόνο για ανθρώπινα δικαιώματα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, δικαιώματα στην ιδιοκτησία κτλ. Από μόνο του είναι ε, κάτι το τελείως ευάλωτο. Το ίδιο θα κάνουμε και για την πολιτική του φίλου, για τις ιδέες ε, τις είπατε, για τα εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολύ ενδιαφέρουσες, πρέπει να το σκεφτούμε, γιατί ε, εγώ έχω αρχίσει να είμαι να έχω επαφές με τα εθνικά κοινοβουλία και ανακαλύπτω πως εμπλέκονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από όσο γνωρίζουμε γιατί κάποιες πολιτικές καθορίζουν το σε τι κόσμο θα ζούμε. Και το θέμα δεν είναι μόνο πόσα λεφτά θα δώσουμε. Αφορά τον κόσμο στον οποίο ζούμε και σε τι κόσμο θέλουμε να ζούμε σε 15-20 χρόνια. αυτή είναι η συζήτηση για την κυρία Στριφλέρ γεωργία, διατροφική ασφάλεια κτλ. θα αποτελέσουν τομέα προτεραιότητας και με τη νέα αυτή πρωτοβουλία για πρώτη φορά έχουμε βάλει ε, υποχρεώσεις ε, για να φέρουμε 7 εκατομμύρια παιδιά να φύγουν από την ένδυα. Και νομίζω πως η μεγαλύτερη πρόκληση για την ανάπτυξη είναι τα υποσυτισμένα παιδιά. Γιατί ξέρουμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και όσο υπάρχει έστω και ένα παιδί που υποσυτίζεται δεν έχουμε κάνει το καθήκον μας. Και πρέπει βεβαίω να εστιάζουμε σε αυτό. Για τον ε, κύριο Σαντιάκο και την διαφοροποίηση. Πράγματι υπάρχουν κάποια σημεία με φτώχεια στην Κίνα. Αλλά αν έχουμε ένα παγκοσμίο πλαίσιο και η Κίνα κάνει αυτά τα οποία αυτά για τα οποία έχει δεσμευτεί, νομίζω πως έχει δυνατότητα να καταπολεμήσει τη φτώχεια. Νομίζω πως το πλαίσιο αυτό του 2015 θα πρέπει να είναι γενικό και εάν αυτή η χώρα καταβάλει προσπάθεια και στο εσωτερικό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αλλά δεν θα βάζουμε εμείς πραγματάκια από εδώ και από εκεί για να ασχοληθούμε με την Κίνα. Δεν επαρκούν κιόλα. και θεωρώ πως πρέπει να είναι ευρύτερη ατζέντα. Για την κυρία Καστίγιο για τις χώρες μέσου εισοδήματο. Χρειαζόμαστε κριτήρια. Πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και ο Τσάρλς ο ίδιος ξεκίνησε αυτή την διαδικασία. Έχουμε και τα μέτρα τα συνοδευτικά της ε, μπανάνας, αλλά το θέμα είναι ποια είναι τα κριτήρια τα οποία έχουμε, γιατί για πρώτη φορά είναι σαφές πως το Κοινοβούλιο θέλει κάποια κριτήρια και αυτό πρέπει να κάνουμε. Αρκεί το ΑΕΠ είναι προσυζήτηση. Αλλά νομίζω πως έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση για αυτά τα οποία είπε η Κριστίνα Γιολάν. Συνεργαζόμαστε καλά με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Θα έλεγα πως έχουμε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι στο παρελθόν. Βελτιώνεται συνεχώς και αναπτύσσουμε μια στρατηγική από κοινού. Για την ερώτηση του κυρίου Φερέιρα. Ε, οι δεσμεύσει βεβαίω πρέπει να εκπληρώνονται και η σημαντικότερη δέσμευση που έχουμε κάνει είναι το 0,7% του ΑΕΠ για την ανάπτυξη μέχρι το 2015. Και είναι σημαντική όθηση του Κοινοβουλίου, ειδικά τώρα που μιλάμε για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ό,τι βάζουμε λοιπόν στον προϋπολογισμό είναι μέρος του 0,7, ένα κρίσιμο μέρος του και θα τελειώσω με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σκέλη για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Νομίζω πως ε, δικαιολογείται. Εγώ είμαι λετονός και ε, μας ενθαρρύνατε πάρα πολύ στη χώρα μου για την ειρήνη, τη σταθερότητα ε, και κάποια ευημερία. Νομίζω πως αυτά είναι αρκετά λόγω της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτές ήταν αλλαγέ που δεν θα ήταν δυνατό να γίνουν με άλλο τρόπο. Και οπωσδήποτε η εμπειρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που πρέπει να προωθήσουμε σε πολλέ περιφέρειε. Σε πολλέ περιοχέ, ειδικά στην Αφρική, όπου πολλέ χώρε μικρέ, αλλά και, η και η Νότιο Αφρική, ε, είναι, είναι αρκετά μικρή. Οπότε ο μόνο τρόπο για να αναπτυχθεί η Αφρική είναι μέσω τη συνεργασία και αποτελεί καλό παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ναι, κύριε Μπρόνς, δεν στηρίζουμε ε, χώρες οπωσδήποτε, προσπαθούμε μέσω των χώρων να εργαστούμε, αλλά στηρίζουμε ανθρώπους. Δεν πρέπει να υπάρχει παρεξήγηση. Ξέρουμε πως βεβαίως ο πιο μόνιμος τρόπος είναι μέσω χωρών ε, και στρατηγικών. Αλλά κάνουμε συχνά την διάκριση ότι στηρίζουμε ανθρώπους. Επίσης για τις χώρες ΑΚΕ Έχουμε τη Συμφωνία Κοτονού μέχρι το 2020. Έχουμε κάποιες δεσμεύσεις, έχουμε διάλογο με τις χώρες ΑΚΕ και ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των χωρών αυτών. Δεν κάνουμε μονομερείς κινήσεις ε, όσον αφορά τη φύση αυτής της σχέσης και ταυτόχρονα θα πρέπει βεβαίως να να συζητιέται και στο Ευρωκοινοβούλιο το τι θα ακολουθήσει την ε, Συμφωνία Κοτονού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από τόσα συγχαρητήρια κύριε Γκέρενς, έχετε τρία λεπτά για να ανακεφαλαιώσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρά τους επένους εγώ θα παραμείνω ταπεινός. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για το ότι εκτίμησαν τη δουλειά που κάναμε στην Επιτροπή. Ξέρω ότι δεν έγιναν δεκτά όλα, ε, όπως η αντίληψη πούμε, της διαφοροποίησης και μιλάμε εδώ για όλες τις γλώσσες της Ένωσης και για όλες ε, τις ε, σημασίες. Έχουμε 112 εκατομμύρια φτωχούς και στην Ευρώπη. Εμείς δεν θα πρέπει όμως να αγνοήσουμε Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τους φτωχούς ανά τον κόσμο και τους φτωχούς ε, στην Ευρώπη, αλλά δεν μπορούμε εμείς να βάζουμε φτωχούς ε, εναντίον φτωχών. Η πολιτική μας της ε, συνεργασίας δεν πρέπει να είναι ούτε αγγελική, ούτε δειλή πρέπει να είναι συνεκτική, αηφόρα. Εγώ εκφράζω την ικανοποίησή μου από αυτήν τη συζήτηση για ορισμένα πράγματα, αλλά έχω και πολλές ερωτήσεις και έχω ένα τεράστιο ερωτηματικό για το αν θα υλοποιήσουμε αυτό το 0,7% δημόσιας βοήθειες μέχρι το 2015. Ο καιρός είναι δύσκολος. Δεν πρέπει να σταματήσουμε να περιφρουρούμε και να, να επαγρυπνούμε συγγνώμη, και να καταβάλουμε τις σωστές προσπάθειες και αν δεν το κάνουμε εμείς κανένας θα το κάνει στη θέση μας θα πρέπει να πληροφορήσουμε καλύτερα και τους πολίτες μας και οι λόγοι ικανοποίησης έχουν να κάνουν με τις απαντήσεις του Επιτρόπου όπου φαίνεται το 2015 να έχει οριστεί ως έτος για την αϊφόρο ανάπτυξη. Αν αυτή η ιδέα ευωδώσει θα πρέπει να δηλώσουμε το 2015 αυτό το οποίο είναι ουσιαστικό για μας στην αναπτυξιακή πολιτική. Δηλαδή η ισχυρή συνεργασία. Ο υπόλοιπος κόσμος αναπτύσσεται ηλικιωδώς. Η Ευρώπη όμως συνεχίζει να έχει βαρύτητα. Εμείς έχουμε μια τεράστια εμπειρία, μια τεράστια τεχνογνωσία, ας κοιτάξουμε να την, πασά, να την περάσουμε στους άλλους, στους συμπολίτε μας και στον υπόλοιπο κόσμο. Επισκέφτηκα πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ευρώπη είναι ο πρώτος χορηγός και η Ευρώπη είναι αντιστρόφως ανάλογη η, ιδέα, η εικόνα της Ευρώπης εκεί και η γνώση για την Ευρώπη είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη βοήθεια που γίνεται. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε με αυτήν την ε, συγκράτηση και ντροπαλοσύνη που δεν αξίζει τον κόπο. Ευχαριστώ. Τελείωσε άρα κοινή συζήτηση. Η ψηφοφορία αύριο στις 6 ώρα. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη οι δηλώσεις του ενός